Uh, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τώρα. Από εκεί, δηλαδή, θα πρέπει να συνεχίσουμε με το υπαριθμό 20 ανακοινώσει του Πρόεδρου. Όμως, οι συντονιστές έλαβαν πολλές αποφάσεις σχετικά με ονόματα εισηγητών κλπ. Και βεβαίως θα σας κοινοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προχωρούμε ε, ε, αμέσως στο 21 που είναι η μελέτη του EPRS της μονάδας δηλαδή εκτονιστέρων των αναλύσεων επιπτώσεων σε θέματα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων την σχετική παρουσίαση θα κάνει η κυρία Εμμανουέλα Τρούλη, λέκτορ στο Τμήμα Οργανώσεως και Δικής Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε στην ε, Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας δίνομαι ευθύς αμέσως το λόγο. Good afternoon. Καλησπέρα σας. Όπως ε, ήδη είπατε, θα κάνω μία παρουσίαση για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διαιρέσεις Η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιο είναι το καθεστώς το οποίο ισχύει σε σχέση με την οδηγία για τις εσωτερικές διαιρέσεις και τη CBND για τις διασυνοριακές. Θα ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση της CBND. Πριν από την θέση σε εφαρμογή του CBND, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις ήταν περίπλοκες και κοστοβόρες και μερικές φορές ήταν απίθαν, αδύνατες σε ορισμένες χώρες. Εναρμονίστηκαν όμως οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το βλέπουμε αυτό με την αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών που έφτασε το 170%. Σχετικά με το περιεχόμενο απαιτείται από όλες τις χώρες της Ένωσης και του Οικονομικού Χώρου να δημιουργήσουν ένα προβλεπτό και ξεκάθαρο, αν θέλετε, πλαίσιο, το οποίο να αυξάνει την λεγόμενη νομική βεβαιότητα, τόσο απαραίτητη για περίπλοκες συναλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, το CBMD διασφαλίζει ότι είναι ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές οι διαμεθοριακές συγχωνεύσεις, προστατεύει τους πιστωτές, επιτυγχάνει συμβασμούς για την προστασία των εργαζομένων, διευκολύνει τις μεταφορές εδρών διαμεθοριακά, επιτυγχάνει κέρδη αποτελεσματικότητας σε ε, σχέση με την αναδιοργάνωση και οδηγεί και σε ε, εξοικονόμηση κόστους. Καθώς συνεχίζουμε την αξιολόγηση του CBMD, ιδίω βλέπουμε ότι διευκόλυνε, αμυσχολείται είναι η ίδια διαφάνεια λέει η κυρία Τρούλη, Προχωρώ στην επόμενη λοιπόν. Παρά όμως τις θετικές ε, πτυχές υπάρχουν και ορισμένα εμπόδια για την πλήρη ανάπτυξη του CBMD. Προβλήματα στην εφαρμογή του CBMD αναφέρονται σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του πλαισίου του και ιδίω το γεγονό ότι καλύπτει μόνο εταιρείε περιορισμένη ευθύνη και μόνο ε, εταιρείε οι οποίες μπορούν να υπό το εθνικό δίκαιο. Η δε προστασία των ε, ενδιαφερομένων μερών, πιστωτών, ε, μειοψηφούντων κλπ. έχει ορισμένα πρακτικά εμπόδια. Πρακτικά εμπόδια που σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή του CBMD, δηλαδή όπω είπα πριν, περιορίζεται μόνο στι εταιρείε ε, περιορισμένη ευθύνη και αυτό μπορεί να είναι αντιφατικό με τον αρχικό του στόχο και σε ό,τι αφορά το άρθρο 1, η οδηγία αναφέρεται μονάχα σε ΕΠΕ που έχουν ιδρυθεί σε συμμόρφωση με το εθνικό δίκαιο. Άρα όχι σε εταιρείες οι οποίες έχουν ε, ιδρυθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έρχονται να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο εμπόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 4.1, οι διαμεθορικές συγχωνεύσεις είναι δυνατές μόνο ανάμεσα σε εταιρείε οι οποίες προκύπτουν από το εθνικό δίκαιο της ε, οικίας χώρας μέλους. Το γεγονό ότι η χώρα μέλος έχει τη δυνατότητα να αποκλείει συγχωνεύσεις ορισμένων εταιριών μεταξύ των, οδηγεί σε φραγμούς στην εφαρμογή των συγχωνεύσεων. Συνεχίζω τώρα με την αξιολόγηση του CBMD. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σχέση και με την προστασία διαφόρων ενδιαφερομένων ε, μερών, για παράδειγμα των μετόχων. Υπάρχει σημαντική απόκληση ανάμεσα στις χώρες, μέλη σε ό,τι αφορά το χρονικό σημείο έναρξης της προστασίας καθώς και στη διάρκεια της. Τις διαδικασίες Υπάρχουν επίσης προβλήματα σχετικά με την προστασία των ε, μειοψηφιών, καθώς και περιπλοκότητες ό,τι αφορά την, ε, την εφαρμογή εθνικών διατάξεων για τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρεία για τον περιορισμό των ε, δικαιωμάτων των μετοχών υπό το νέο εθνικό καθεστώς, καθώς και την πληρωμή αποζημιώσεων στους μειοψηφούτες μετόχους. Όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Στο CMDMD προτείνονται κάποιες λύσεις που οδηγούν σε κάποιες εύθραυστες συμβιβαστικές λύσεις. Υπάρχουν όμως και κάποια, θα έλεγα, διφορούμενα θέματα, στα οποία θα μπορούσε να απαιτηθεί περισσότερη διευκρίνηση. Για θέματα τα οποία αφορούν τα δικονομικά και προπτικά προβλήματα, έχουν υπάρξει θέματα στον τομέα της τεκμηρίωσης, οι διαδικασίες fast track σε περιπτώσεις ταχείας αναδιοργάνωσης φυγατρικών και κύριων εταιριών. όπως επίσης και προβλήματα σχετικά με την έναρξη και τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Um, uh, Αποτίμησης. Σχετικά τώρα με τις εσωτερικές διαιρέσεις και όχι οι διαμεθοριακές. Καλύπτεται η κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών σε εθνικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο διαμεθοριακό. Οι διασπάσεις λοιπόν εφαρμόζεται σε κράτη-μέλη ε, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία παρά την έλλειψη, αν θέλετε, κάποιων συγκεκριμένων ρυθμίσεων, υποχρεωτικών και δεσμευτικών, υπάρχουν μηχανισμοί εθνικοί που επιτρέπουν τις διασυνοριακές διαιρέσεις ή διασπάσεις. Διευρύνεται δηλαδή η εμβέλεια το πεδίο εφαρμογής του CBMD μέσω του λεγόμενου gold plating και σε μια διαφορετική κατηγορία χωρών η νομοθεσία που να επιτρέπει για τέτοιου είδους διασπάσεις υπάρχει ανεξαρτήτως της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία του CBMD. Αλλά σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν καθόλου τέτοιου είδους δυνατότητες. Συνολικά λοιπόν υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη σχετικά με τις διασυνοριακές τέτοιου είδους διαιρέσεις. Σχετικά λοιπόν με την οδηγία για τις εσωτερικές διασπάσεις <clears throat> υπάρχει έλλειψη αν θέλετε νομικής βεβαιότητας σε σχέση με τις επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης η μη ύπαρξη μιας διαρθρωμένης διαδικασίας για τις διασύνοριακές διαιρέσεις είναι σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα, μηχανισμοί που θα επιτρέπουν αυτού του είδους τις διασπάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενημέρωσε, δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο το 2015 και λέγει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι συμβαλόμενοι είναι υπέρ της δημιουργίας ενιαίας νομοθεσίας. Η πρόταση κωδικοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ουσία ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό κείμενο τις προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν ήδη και στη CBMD και στην οδηγία για εσωτερικές διασπάσεις. Πρόκειται για μια κωδικοποιητική διαδικασία που δεν εισάγει τίποτα το καινούριο σε σχέση με τις διασυνοριακές διαιρέσεις και το, στην, την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα αυτό. Σχετικά τώρα με τις δυνατότητες βελτίωσης, το θέμα είναι πώς οι βελτιώσεις αυτές θα υπάρξουν σαν παράδειγμα προτάσεις για την προστασία των πισωστών και των μετόχων. Πλήρης εναρμόνιση είναι η πρώτη επιλογή. Συγκεκριμένο, αν θέλετε, ε, συγκεκριμένος κατάλογος μέτρων, το δεύτερο και ανοιχτός κατάλογος μέτρων, το τρίτο, η τρίτη επιλογή καλύτερα. Η τρίτη επιλογή θα βασιστεί στις πιο διαδεδομένες πρακτικές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τα δικαιώματα των μετόχων που μειοψηφούν όπως επίσης και τα δικαιώματα των πιστωτών θα προστατευθούν. Οι δυνατότητες θα είναι ανοιχτές ε, να διαλέξουν τα κράτη-μέλη ή την ε, προστασία της υψηλής κινητικότητας ή την προστασία των μετόχων σαν πρώτο ε, επίπεδο προστασίας. Υπάρχει η δυνατότητα λοιπόν επίσης ανάμιξης διαφορετικών επιλογών αυτό θα δώσει στα κράτη-μέλη υψηλό επίπεδο διακριτικής, αν θέλετε, δυνατότητας λύσης των προβλημάτων ε, και σίγουρα όμως περιορίζει τα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουν ε, τα κράτη-μέλη. Σχετικά με τα συμπεράσματα τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το CBMD είναι ένα πετυχημένο μέσο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εμπόδια στην πλήρη αποτελεσματικότητά του. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να ξεπεραστούν μέσω μιας αναθεώρησης του CBMD που να αντιμετωπίζει κάποια από τα εξή θέματα. Διεύρυνση της εμβέλειας του CBMD για όλα τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 54 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης. Περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων για την προστασία των πιστωτών, πιθανώς με την εισαγωγή ε, και ενός συστήματος προστασίας εκ των υστέρων που δεν θα καθυστερεί τη συγχώνευση εναρμόνιση επίσης της προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων, κατάλληλη αποζημίωση και συμπληρωματική αποζημίωση σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ε, βίαιη ή μη κατάλληλη αν θέλετε αλλαγή του λόγου ε, ανταλλαγής των μετοχών. Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις ε, της έκθεσης για τη συγχώνευση, ε, συμμετοχή και καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στις εθνικές αρχές, προσεκτικές ρυθμίσεις για την προστασία επίσης των κανόνων που διέπουν μάλλον την προστασία των εργαζομένων. Σχετικά τώρα με τις ε, διασπάσεις ε, πέραν τις διασυνοριακές. Η οδηγία η οποία αυτή τη στιγμή είναι πλήρως ενισχύει καλύπτει μόνο τις εσωτερικές διασπάσεις. Η σημερινή κατάσταση δίνει την δυνατότητα μόνο σε ορισμένες χώρες να έχουν ξεκινήσει τέτοιου διαδικασίες, τέτοιου είδους διαδικασίες και οι υπόλοιπες χώρες χρησιμοποιούν πάρα, πολλά, πάρα πολύ περίπλοκες διαδικασίες και μέτρα, κάτι το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση διόλου ικανοποιητική που απαγορεύει ουσιαστικά σε ορισμένες περιπτώσεις την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και παραβιάζει και το δικαίωμα της ελευθερίας εγκατάστασης. Ένα νέο πλαίσιο λοιπόν για τις διασυνοριακές διασπάσεις θα πρέπει να προταθεί σε σχέση πάντα με τις προτάσεις για το CBMD, τα μέλη του Κοινοβουλίου δικαιολογημένα έχουν ενδιαφερθεί για τους τρόπους διευκόλυνσης της κινητικότητας των επιχειρήσεων είτε μέσω της αναθεώρησης του CBMD είτε δημιουργώντας νέους κανόνες για τις διασυνοριακές διασπάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ κυρία μου και για την παρουσίασή σας και την παρουσία σας. Και τώρα η σειρά των ε, Ευρωβουλευτών να σχολιάσουν ή να κάνουν ερωτήσεις, εάν το επιθυμούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως και την ε, κυρία Τρούλη για την παρέμβασή της και τις πολλές εξηγήσεις που έδωσε. Ωστόσο αυτές ήταν κάπως θεωρητικές, αν μπορεί να τους εμφυσίσει κάποια ζωή να μας δώσει δηλαδή μια συνολικότερη επισκόπηση για πόσες συγχωνεύσεις ή διασπάσεις μιλούμε ένα έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες πλήττονται εντό εισαγωγικών περισσότερο ή άλλες λιγότερο. Και όταν λέτε ότι υπάρχουν ακόμα κολλήματα, εμπόδια, φραγμοί στις συγχωνεύσεις αλλά και στις διασπάσεις, μήπως μπορείτε να μας δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα όταν θέλουν για παράδειγμα να συγχωνευτούν δύο επιχειρήσεις. Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να με βοηθήσετε να αντιμετωπίσω και τα θέματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης. Αν είναι δυνατόν να μας δώσετε λίγα συγκεκριμένα παραδείγματα από την πρακτική για να δούμε πού εντοπίζονται τα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις απαντήσεις που θα δώσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω, λέει ο πρόεδρος πλέον, άλλον που να επιθυμεί να λάβει το λόγο. Μπορώ λοιπόν να επιστρέψω το μικρόφωνο στην κυρία Τρούλη. Μου επιτρέπετε να ερωτήσω. Η ερώτησή σας αναφέρεται στο status quo ante πριν από το CBMT ή στην ε, νυν κατάσταση. Υπάρχουν αναφορές στην έκθεσή μας με πολλά διαφορετικά παραδείγματα. Έχουμε μια μελέτη περιπτώσεως, μια case study. Υπάρχουν διαφορετικά παραδείγματα σε σχέση με κάθε είδους κόλλημα που έχουμε διαπιστώσει. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής, αναφερόμαστε σε σχηματισμούς, σε συγχωνεύσεις που δεν μπορούν να γίνουν τελικά, δίνουμε και παραδείγματα, περιπτώσεων που δεν καλύπτει το τρέχον πεδίο εφαρμογή του CBMD. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων εκεί, επίσης έχουμε παραδείγματα. Ε, δεν είμαι βέβαια αν θέλετε ένα... Αν έχετε κάτι που σας ενδιαφέρει συγκεκριμένα. Έχω μια μικρή περίπτωση εδώ. Η παριθμόν 45 τις λογιστικές επιπτώσεις της εφαρμογής της EBMD μεταξύ Γερμανίας και Ρουμανίας, μεταξύ γερμανικών και ρουμανικών εταιριών. Η γερμανική εταιρεία ε, ήταν θεσπισμένη ήδη από πριν, ενώ η ρουμανική για την η συγκεκριμένη ημερομηνία δηλαδή ε, δημιουργία της είναι και υπάρχει μια διαφορά. Εάν τώρα θέλει η γερμανική εταιρεία να συμφωνηθεί με τη ρουμανική εταιρεία, εκεί θα υπάρχει ένα κενό χρονικό. Και αντίθετα, εάν η ρουμανική επιχείρηση θέλει να συγχωνευτεί στην γερμανική, θα υπάρξει το πρόβλημα από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, θα πρέπει να βάλει σε λογιστικές μονάδες τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της η ρουμανική εταιρεία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εφόσον έχετε ενδιαφέρον για κάποιο ιδιαίτερο θέμα, δεν θέλω να σα φορτώσω περισσότερο, αλλά ε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μπορώ να σας ε, παρουσιάσω. Άλλος κανείς? Δεν έχω άλλο κανένα. Σας ευχαριστώ, ε, Δόκτωρ Τρούλη, και πάλι για την παρουσίαση. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι σε ένα βαθμό παρόμοιο εξέταση σχεδίου εκθέσεως για διαμεθοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Τον λόγο λαμβάνει ο κύριος Γκασμπάρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Τρούλη για την μελέτη που έκανε. Θα την κοιτάξω τη μελέτη αυτή με μεγαλύτερη προσοχή βεβαίως, αλλά νομίζω ότι προκύπτει από αυτά που μας είπε σήμερα μία ανάλυση την οποία συμμεριζόμαστε και ούτως ή άλλως έχω συμπεριλάβει και στην πρότασή μου στην πρόταση έκθεσης. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που έχει η ισχύουσα οδηγία, η οποία οδηγία έχει και θετικές πτυχές, προφανώς γιατί διευκόλυνε πολλές διασυνοριακές λειτουργίες, μείωσε πάρα πολύ το κόστος των διαφόρων επιχειρήσεων και έδωσε νέα δυναμικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο. Αλλά προφανώς τώρα μετά από πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μετά από τις πολλές δυσκολίε που έχουμε γνωρίσει και τα παραδείγματα που μας αναφέρθηκαν και που αναφέρει και η μελέτη και τα οποία θα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά σε ό,τι αφορά προβλήματα σε σχέση με τις συγχωνεύσεις, αλλά κυρίως το πρόβλημα που απορρέει από την έλλειψη μιας συγκεκριμένης οδηγίας για τις διασπάσεις των επιχειρήσεων Νομίζω λοιπόν ότι μετά από όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει, καλό θα ήταν να ετοιμάσουμε μία έκθεση όπου θα υπάρχει, πάνω γύρω από την οποία θα υπάρχει βρία συνένεση πριν από το καλοκαίρι, πριν από την ολομέλεια, τελευταία ολομέλεια του καλοκαιριού, ούτως ώστε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ετοιμάζει την νομοθετική μεταρρύθμιση της οδηγίας για το συγκεκριμένο θέμα, να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να βάλει τις απαραίτητες αλλαγές, να κάνει όλες αυτές τις τροποποιήσεις μετά από την εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει τα τελευταία δέκα χρόνια ε, για το τι επιπτώσεις είχε η οδηγία στις επιχειρήσεις, στο, στους εργαζομένους κτλ. Και, ε, και να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις εξέλιξεις και αυτή την εμπειρία. Η πρόταση που κάνω εγώ σήμερα είναι μια ανοιχτή πρόταση. Παρουσιάζω στους συναδέλφους κάποιες ιδέες και ζητάω τη συνεισφορά όλων σε αυτή την προσπάθεια. Από σήμερα μέχρι την τελική έγκριση αυτού του κειμένου. Και βασίζομαι, βασίζομαι σε δύο άξονες. Καταρχάς, το γεγονός ότι θα αναθεωρήσουμε την οδηγία για τις συγχωνεύσεις, εντάξει, από τη μία είναι αυτό, και από την άλλη θα πρέπει να προβλέψουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση ε, σε θέματα διακυβέρνησης των, ε, των επιχειρήσεων ε, και τι, πώς προστατεύουμε τα, τους μειοψηφούντες μετόχους. Και επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν επιπτώσεις στην ταμιακή νομοθεσία, ξεκάθαροι ορισμοί των τυποποιημένων εγγράφων κτλ, εναρμόνιση των κανόνων, στα εξή θέματα. Διαχείριση των επιχειρήσεων, μέθοδο της αξιολόγηση της δραστηριότητα και αποτίμηση, αρχή και διάρκεια της περίοδου προστασίας για τους πιστωτέ με βάση την αρχή ε, των ευθυνών που προκύπτει από την ε, Γενική Συνέλευση, ε, καλύτερη προστασία των ε, μειοψηφούν των μετόχων, έρευνα στους, στις συγχωνεύσεις, ε, αποζημιώσεις σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφισβήτηση. Φυσικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, εξαιρεσει και επιταχυμένε διαδικασίες σε περιπτώσεις που υπάρχει σαφέστατη συνένεση. Τέλος, σε σχέση με τους ισχύοντε κανόνες για το κανονισμό που αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να αποφύγουμε κάποιε επιχειρήσει να χρησιμοποιήσουν την οδηγία για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ε, για να μεταφέρουν την εταιρική έδρα μόνο και μόνο για λόγους φορολογικούς, ε, κοινωνικούς ή νομικούς. Τελευταίο σημείο που αγγίζουμε είναι το σημείο που αφορά τις, ε, τις διασπάσεις. Ελπίζουμε ότι η νομοθετική μεταρρύθμιση της Κομισιόν θα συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή που έλειπε από την ε, οδηγία του 2005, δηλαδή για τις διαστημικές συγχωνεύσει CBMD. Και ελπίζουμε να μπουν ειδικοί κανόνες ε, που απαιτεί η ατυχία, κυρίω για τα δικαιώματα των πιστωτών, ε, τα δικαιώματα των μειοψηφούντων πιστωτών, για την ε, συμμετοχή και την προστασία των εργαζομένων για, και για τις διαδικασίε. διαδικασίες. Σημείο 2, τη ρύθμιση όλων των βασικών περιπτώσεων ε, συγχώνευσης που βλέπουμε σήμερα να υπάρχουν στην αγορά. Η πρότασή μου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε η Κομισιόν και που ολοκληρώθηκε το 2015, δηλαδή σε όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης, όπου συμμετείχαν επαγγελματίες του κλάδου ε, και ειδικοί. Και αν οι συνάδελφοι συμφωνούν, εγώ θα πρότεινα μέχρι να ε, εγκριθεί το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια ε, πριν από το καλοκαίρι, του Ιουλίου δηλαδή, μέχρι τότε να, είμαστε, να αφήσουμε ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα, έτσι, ανοιχτό ας πούμε τον ορίζοντα και μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου να έχουμε περιθώριο για τους συμβασμούς, έτσι, τις, ε, τους συναδέλφους της Επιτροπής Γιούρη και να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γιούρη το Μάιο και να ψηφίσουμε τελικά για το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια πριν το καλοκαίρι. Πριν την καλοκαιρινή, δηλαδή το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κανένα να σχολιάσει. Ποιο ευρωβουλευτή παρακαλώ θα ήθελε να σχολιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, να συγχαρώ τον κύριο Γκασπάρα για την έκθεσή του για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις το εταιρικό δίκαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κινητικότητα των επιχειρήσεων στα πλαίσια της ε, ενίας αγοράς. Η διευκόλυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων αποδείχτηκε πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, απόδειξη είναι ο αυξημένος αριθμό των συγχωνεύσεων από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία. Συμφωνώ ότι οι κανόνε για τι διασυνοριακές ε, συγχωνεύσει ε, θα πρέπει να επανεξεταστούν και να διευκρινιστούν και μέσω της υιοθέτηση νέων πολυ, πολύγλωσσων εντύπων και με την υιοθέτηση νέων πρακτικών ε, χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία, την πληροφορική δηλαδή. Η μεταρρύθμιση της οδηγίας δεν θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να συμπεριλάβουμε και τις διασυνοριακές διασπάσεις, καθώς και την μεταφορά της εταιρική έδρας. Όταν αυτή γίνεται για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την φοροαποφυγή. Ε, πρέπει να εναρμονίσουμε αυτές τις αστυνοριακές έτσι, λειτουργίες, συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μεταφορές εδρών. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα της προστασίας των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Δεδομένης όμως της ε, εξειδικευμένης ε, φύσης ε, του νομοθετήματος αυτού και δεδομένου του, Τη πολιτική ευαισθησία που υπάρχει, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί πάρα πολύ και να μπει στην καρδιά των συζητήσεών μας. Θα πρέπει να το θέσουμε αυτό το θέμα, να το εξετάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συζητάμε και θέματα προστασίας των εργαζομένων και μέσα εκεί να συζητηθεί και αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Άλλος δεν ζητεί τον λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στην διαδικασία επεξεργασίας του προγραμματός μας. Για το λόγο αυτό προτιμούμε να απέχουμε από σχόλια. Καλώς, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο εισηγητής επιθυμεί να λάβει τον λόγο πάλι. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ράντου. Το θέμα της προστασίας των εργαζομένων συμπεριλαμβάνεται. Και φυσικά η προστασία των εργαζομένων δεν αφορά μόνο αυτόν τον τομέα. Το έχει πει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο σε διάφορες φάσεις, σε διάφορες συζητήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω του συναδέλφου αν συμφωνούν με το χρονοδιάγραμμα που, που, έχω πρότεινα. Και η Κομισιόν βεβαίω αν συμφωνεί με αυτό. any... Ο πρόεδρο δεν είδα κανένα γύρι ένσταση. Δεν είδα καμία ένσταση ούτε από τα μέλη ούτε από την γραμματεία. Άρα μου φαίνεται ότι έχει καλώ. Άρα μπορούμε τώρα εδώ να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του θέματος αυτού και να συνεχίσουμε με το υπαριθμό 24 Πρόκειται για την ερμηνεία και υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας για την βελτίωση της νομοθεσίας. Εδώ συνεισηγητής είμαι ο ίδιος προσωπικά. Θα ήθελα λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι στις 26 Ιανουαρίου ενεστώτος έτους η ομάδα εργασίας προχώρησε στην έκτη συνάντησή της με βασικά θέματα στην ημερησία μας διάταξη ανταλλαγή απόψεων με τον Μάρκους Βίνκλερ, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Task Force Γραμματέα του Κοινοβουλίου για τη βελτίωση νομοθεσίας. Δεύτερο, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εμπειρίες διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών όσον αφορά την διαφάνεια και τον συντονισμό της νομοθετικής διαδικασίας μέσα στα πλαίσια πάντα της Διοργανικής Συμφωνίας. Η ομάδα εργασίας άκουσε τον κύριο Βίνκλερ, ο οποίος τόνισε ότι παρόλο που στη Γεωργιανική Συμφωνία έχουν συζητηθεί τα περισσότερες ανάγκες του Ευρωκοινοβουλίου, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά θέματα, όπως η διάκριση μεταξύ κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων ο συνδυασμός τραπεζών δεδομένων για την πρόοδο της εξελίξεως των νομοθετικών φακέλων, όπου εκεί το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει και να επιτύχει περισσότερη διαφάνεια. Τόνισε ακόμη ότι το πιο κρίσιμο σημείο είναι να επιτευθεί η ορθή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διαφάνειας και στην προστασία μιας ζώνης που να διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που ε, μπορούν να θεωρηθούν ορθές. Η Προεδρία απάντησε και στο αίτημα του ε, διαμεσολαβητού για την κοινή δήλωση για τον προγραμματισμό που συνυπογράφουν τα τρία θεσμικά όργανα, για κοινέ συνεδεύσει τύπου και για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το Μητρό Διαφάνειας, μεταξύ άλλων τα μέλη της ομάδας εργασίας τοποθετήθηκαν ή έθεσαν ερωτήσεις για την συνέχιση εργασίας της Task Force για την εφαρμογή της παραγράφου 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για την δημοσίευση εγγράφων που προέρχονται από τριμερείς διαλόγους και για το νέο άρθρο 69 γάμα. για τα κριτήρια οριοθέτησης και για τους μηχανισμούς ενημέρωσης για τους τριμερείς διαλόγους, για τις αξιολογήσεις αντικτύπων στους τριμερείς διαλόγους και για, την, για το ρόλο του Κοινοβουλίου στην πρόθεση της διαφάνειας. Η ομάδα εργασίας άκουσε και τις απόψεις της κυρίας Φόρντ, Προέδρου της Επιτροπής ΙΜΚΟ, καθώς και του Γουαλτιέρη της Επιτροπής ΕΚΟΝ, οι οποίοι ανέπτυξαν τις εμπειρίες τους ό,τι αφορά την διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία. Ιδιαιτέρως η κυρία Φόρντ αναφέρθηκε στους μηχανισμούς που επιτρέπουν υψηλά πρότυπα διαφάνειας στο έργο της Επιτροπής της. Εξέφρασε και τις επιθυμίες της για βελτίωση διαφάνειας και από πλευράς άλλων θεσμικών οργάνων και έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαφάνεια εντός του Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Γκουαλτιέρη αναφέρθηκε στην απομακρού πρακτική της Επιτροπής του και θεωρεί ότι και οι νέες διατάξεις του κανονισμού πρέπει να κινηθούν προς τη διακατεύθυνση. Αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται για, την... για τον συντονισμό των... Ε, του προγραμματισμού εργασιών με το Συμβούλιο και θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο είναι διαφανέστερο του Συμβουλίου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της εκθέσεώς μου. Κανονικά θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην κυρία Χάουταλα, η οποία ήταν παρούσα στη συνάντηση, δυστυχώς ε, δεν είναι παρούσα. Μπορώ λοιπόν να δώσω τον λόγο σε κάποιο από τα μέλη που είναι παρόντα, εφόσον επιθυμούν. Αλλά δεν βλέπω κανέναν να, ε, ε, ε, να ενδιαφέρον. Άρα ολοκληρώνεται εδώ το θέμα αυτό. Α, δεν είναι παρόν και ο είναι. Ο πρόεδρος, έχουμε ένα πρόβλημα διότι για τα κοινά σημεία που είναι τα 25 και 26 δεν είναι παρόν ο κύριος Άντερσον που είναι εισηγητής και για το 28 επίσης μας λείπει ο κύριος Λεμπρετόν Αν συμφωνείτε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να αναζητηθούν τα πρόσωπα αυτά. Πέντε λεπτά αν συμφωνείτε. Okay, so we have Mr. Anderson among ourselves. So... Θα, θα συγχωνεύσουμε κατά κάποιο τρόπο τα σημεία 25 και 26 και έτσι θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Άντερσον. Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την ταχεία ψήφιση και κύρωση του νομοθετικού πακέτου ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συνθήκη. Αυτό είναι και ο ρόλο μα ω Ευρωβουλευτών. Και αυτό είναι βεβαίω ο δικό μου ιδιαίτερο ρόλο ω εισηγητού. Η συνθήκη για την οποία μιλώ ε, ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση με την ε, συμβολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε ταχύτατα και να εγκρίνουμε τις ε, τροπολογίες. Μιλούμε για μια στενή συνεργασία εποφελία ορισμένων κατηγοριών προσώπων που θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν αυτό τον λοιμό βιβλίων, την έλλειψη, την στέρηση βιβλίων για ανθρώπους με ε, συγκεκριμένες αναπηρίες, ε, τυφλούς, αμβλίωπες και με άλλα προβλήματα ανάγνωσης πολύ ευχαρίστως εργάζομαι υπέρ της ε, πρόθεσης και εφαρμογής και κύρωσης της σχετικής ε, συνθήκης μαζί στη συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες επιτροπές, την Επιτροπή Ίντα, Απασχολήσεως, Πολιτισμού και Αναφορών. Όλες οι επιτροπές αυτές επιθυμούν να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν η έγκριση των ε, ε, προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ επίσης. ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε πει να ψηφίσουμε σήμερα. Όμως δεχθήκαμε να αναβάλουμε για ένα μήνα, τέλη Φεβρουαρίου, ώστε να δώσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα κείμενα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, άλλε επιτροπέ έχουν ήδη εγκρίνει γνωμοδοτήσεις τους. Επειδή πρόκειται για σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο χρειάζεται ταχεία εφαρμογή, θα μπορέσουμε, πιστεύουμε, να ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο, διότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτές είναι σύμφωνοι. Υπάρχουν σχεδόν 100 τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Έχοντας διαβάσει όλες τις τροπολογίες αυτές, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ευρύς ε, συμβιβασμούς και μάλιστα πολύ σύντομα. Thank Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Επιθυμεί άλλο μέλος ε, της Επιτροπής. Εσείς κύριε Νεγκρέσκου. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη συνεργασία. η έκθεση θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να εμείνουμε στο πεδίο εφαρμογής. Είναι σημαντική έκθεση ε, διότι θα μπορέσει έτσι να εξυπηρετήσει τους τυφλούς και ελπίζω το Συμβούλιο να ακούσει τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βεβαίως και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο. Νομίζω ότι όλοι οι παρόντες συμμερίζονται την άποψη την οποία εξέφρασε ο κύριος Νεκρέσκου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε τη δυνατότητα χθες σε μια πιο ανεπίσημη συνάντηση να μεταφέρουμε τις απόψεις μας και τα αισθήματά μας για την πρόταση αυτή. Εμείς είμαστε υπέρ της άποψης που εκφράζει το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια γρήγορη και ήρεμη διαδικασία αποδοχής αυτών των δύο προτάσεων και γενικότερα πιστεύουμε ότι και το Συμβούλιο συμφωνεί με μας έτσι ώστε να υπάρξει σε έλογο χρονικό διάστημα μια σωστή λύση. Είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν από τις προτάσεις και περιμένουμε τα επόμενα στάδια, τις επόμενες φάσεις. Okay. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι και η Προεδρία σημείωσε τη σημασία που δίνουμε εμείς στα δύο αυτά θέματα. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από πλευρά Συμβουλίου, δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν χρόνος υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο και γι' αυτό θα κλείσουμε τα δύο αυτά τα θέματα. Έχουμε ένα θέμα μπροστά μας προς συζήτηση μόνον. Ο εισηγητής του θέματος αυτού, ο κύριος Λεμπρετό, έρχεται, θα φτάσει σε πέντε λεπτά, οπότε για μια ακόμη φορά ε, θα του δώσουμε την δυνατότητα να εκφραστεί στην μορφή γλώσσα του Μολιέρου. Dear colleagues, we may continue. Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε. Με το άρθρο 28, εξέταση πρότασης γνωμοδότησης για την προστασία απέναντι σε προϊόντα ε, dumping και επιδοτήσεων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Λεμπρετό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στόχος αυτής της πρότασης είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 1036 και 1037 εναντίον του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων. Το πρωτόκολλο συνεργασίας της Κίνας με τον ΠΟΕ ε, τελειώνει σε λίγους μήνες και μιας και η Κίνα θέλει να πάρει το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς, θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενε αλλαγές. Μέχρι τώρα, για να δούμε αν υπάρχει κίνδυνος dumping, συγκρίναμε ένα εξαγόμενο προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την τιμή του προϊόντος σε μία αντίστοιχη με την Κίνα χώρα, όπως η Βραζιλία. Μετά από την σύγκριση αυτή, μπορούσαμε να καθορίσουμε το ύψος των ε, δασμών. Το σύστημα αυτό δεν θα συνεχιστεί μετά από αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου και γι' αυτό προβλέπεται ένα νέο σύστημα το οποίο θα δίνει κατά τομέα συγκεκριμένες μελέτες για τις τιμές στην Κίνα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και την δυνατότητα συνέχισης του προηγούμενου συστήματος με τέλη δηλαδή αντίστοιχα στην περίπτωση που υπάρχει σημαντική στρέβλωση στην αγορά. Είναι μια πρόταση που δεν ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δημιουργεί πάρα πολλούς φόβους, διότι το βάρος της απόδειξης είναι από την πλευρά των Ευρωπαίων. Ενώ στην περίπτωση όπου υπάρχουν αμφιβολίες, η Κίνα θα πρέπει να είναι αυτή που θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει dumping. Μιλάμε για ένα σύστημα λοιπόν ανεπαρκώς προστατευόμενο και γι' αυτό ζητάμε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να απορρίψει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα επιχείρηματα του εισηγητή ε, άκουσα δηλαδή τον λόγο για τον οποίο προτείνει την απόρριψη της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ αντίθετα θεωρώ ότι κάτω από τις ισχύουσες νέες πλέον συνθήκες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε πράγματι την ευρωπαϊκή οικονομία. Βλέπουμε τι κάνουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει αντίστοιχα με τους Αμερικανούς μέτρα γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες είναι καθοριστικές για τις οικονομίες μας και οι εισαγωγές που φτάνουν στις ευρωπαϊκές αγορές απειλούν τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Συνεπώς, εγώ είμαι υπέρ της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί τα μέσα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξισορροπούν σωστά τα συμφέροντά μας για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ακριβώς τα συγκεκριμένα συμφέροντα από το dumping άλλων χωρών. Μη μελών. Θυμίζω ότι η σημερινή κατάσταση μας υποχρεώνει να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματικοί, γιατί αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι θα μείνουμε γενικά εκτός. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. Θα ζητούσα κανονικά από την Κομισιόν να πάρει το λόγο, αλλά δεν εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή. Σημειώστε τότε ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Δευτέρα, 6 ε, Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα. Δεν έχετε αντιρρήσεις, αν δεν έχετε. Προχωράμε εκτός και αν θέλει ο εισηγητής να αντιδράσει στο σχολείο του κυρίου Μπούντα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούντα που εξέφρασε την άποψή του. Συμφωνούμε επί της αρχής. Δηλαδή ότι πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία εναντίον πιθανότητα της απόπειρας dumping από το εξωτερικό. Αλλά φυσικά εκτιμούμε με τελείως διαφορετικό τρόπο τις λύσεις που πρέπει να πάρουμε. Εγώ προτείνω την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν, όχι γιατί ε, είναι εντελώ κακή, αλλά γιατί είναι ανεπαρκή. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα καλύτερα μέτρα, πιο προστατευτικά. Περί αυτού πρόκειται. Η διαφορά δεν είναι στο πώς ριζική, ας πούμε, σε απόψεις μας, αλλά είναι διαφορά βαθμού. Πώς εκτιμούμε την προστασία, δηλαδή, που εξασφαλίζει η πρόταση. Μια και έχουμε χρόνο να αντιδράσω, Πρόεδρε. Υπάρχουν προτάσει από πλευρά Κομισιόν μερικέ φορέ που δεν πάνε αρκετά μακριά. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι να απορρίψουμε την πρόταση. Νομίζω αντίθετα ότι η λύση βρίσκεται στο να την τροποποιήσουμε την πρόταση αυτή τη Κομισιόν. Ούτω ώστε να υλοποιεί του στόχου που επιθυμούμε όλοι. Την προστασία δηλαδή των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν απορρίψουμε την πρόταση, θα έχουμε καθυστερήσει, θα επιστρέψει το θέμα στο γήπεδο της Κομισιόν και σας λέω ακόμα μια φορά, ξυπνήστε. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό και πρέπει να αντιδρούμε εγκαίρω, όχι με μεγάλη καθυστέρηση. Γι' αυτό τροποποιήστε την πρόταση, αλλά μην την απορρίψετε. Τότε περιμένω τις ε, τροπολογίες σας με μεγάλο ενδιαφέρον. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Το μόνο που θέλω να πω λοιπόν για αυτό το σημείο και με αυτό κλείνω είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει στις Βρυξέλλες, Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου, από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Κλείνουμε με αυτό το σημείο την ημερήσια διάταξη και σας ευχαριστώ που ε, ήρθατε εδώ.